για να εξισορροπήσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θέλει να υποστηρίξει τη δημόσια επένδυση, αλλά εμεί θέλουμε να το στρέψουμε περισσότερο στη στήριξη της ζήτησης και όχι της προσφοράς. Και ένα ε, σύστημα Αλλά ε, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και ο κύριος Μπέκ αγορές και προς τα έξω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έμαθε από τις κρίσεις και κινητοποιεί ή ε, ε, στείνει εργαλεία για να αντιμετωπίσει την επόμενη κρίση, η οποία θα έρθει. Δεν ξέρουμε πότε, αλλά θα τη βρούμε μπροστά μας και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αργούμε λίγο γιατί το καλό το πράγμα αργεί να γίνει, αλλά αντιδρούμε, εν πάση περιπτώσει ποιο είναι το εκ των όνων κάνευ, να είναι αυτόματος ο σταθεροποιητής. Αν δεν μπει αυτόματος χαρακτήρας, δεν θα έχει την ε, αποτελεσματικότητα που οφείλει. Και το χειρότερο ποιο είναι, 30 δις για όλη την Ευρωζώνη, καλά, σιγά τα λεφτά, ούτε έχει και τεράστιο αντίκτυπο, αλλά μπορεί να αυξηθεί η πρόταση. Ένα μικρό δημοσιονομικό σχόλιο. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το, ε, το μέσο αυτό είναι εκτός ε, των οροφών του δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά θα πρέπει να εντάσσεται στην οροφή των ιδίων πόρων. Όταν ορίσουμε τις ποσότητες και τα ποσά μάλλον, δεν θα πρέπει να μειωθεί το PDP, καλύτερο είναι αυτοματοποίηση, το χειρότερο είναι το ποσόν και αυτό που λείπει και συμφωνώ με τα όσα έλεγε προηγουμένως η κυρία Μπερές είναι η ασφάλεια της ανεργίας. Για πρώτη φορά την ασφάλεια και αντασφάλιση της ανεργίας. Όλο και περισσότερες χώρες το βλέπουν αυτό ευνοϊκά και το Κοινοβούλιο θα διέπρεται μέγα σφάλμα εάν δεν τα έβαζε αυτά στο συγκεκριμένο κανονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Μουρεσάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα συνάδελφοι. Σε πρώτη φάση θέλω εκ μέρου τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να ευχαριστήσω του δύο συνεισηγητέ, Μπερέ Μπέγκε, για την δουλειά του που δεν έχει σταματήσει και που ξεκίνησε από πέρσι με την δημοσιονομική δυνατότητα της ε, Ευρωζώνης που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο. Κατά πρώτον να πω ότι εκτιμώ το γεγονός ότι οι συνάδελφοι ρητός καλούν στην έκθεση για τακτική υποβολή εκθέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο σε σχέση με την εξέλιξη του μηχανισμού αυτό θα πρέπει να το επιδιώξουμε. Έναν ισχυρότερο ρόλο του Κοινοβουλίου σε όλο αυτό το νέο σχήμα. Επίσης, ε, συμφωνώ με την αιρεσιμότητα. Η αιρεσιμότητα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, να είναι μικροοικονομική, να είναι μικροοικονομικά τα κριτήρια δηλαδή και με περισσότερο να δώσουμε και τις λεπτομέρειες. Υπάρχει εδώ και ένα σημαντικό πολιτικό στοιχείο Δηλαδή, η αιρεσιμότητα θα πρέπει να έχει να κάνει με το σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών και το κράτο δικαίου και να μην ε, μπορεί να βοηθηθεί μια χώρα που είναι στη δικασία του άρθρου 7. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Είναι ένα στοιχείο άκρο πολιτικό και θα πρέπει να σκεφτούμε τι επόμενε εβδομάδε αν θα το προκρίνουμε ή όχι. Ε, πέραν αυτών, ήθελα να επιμείνω σε κάποια σημεία που θα ήθελα να το αναλύσουμε καλύτερα με του συναδέλφου και του εισηγητέ και χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα θέμα σύγκλησης. Ένα κώδικα μάλλον σύγκληση, ο οποίο καλό είναι να υπάρχει. Την καλωσορίζω την ιδέα, αλλά δεν θέλουμε να αντικαταστήσει την υπάρχουσα δημοσιονομική νομοθεσία. νομοθεσία. Θα πρέπει να είναι κάτι το πρόσθετο σεβασμό του κώδικα αυτού σε σχέση με του κανόνε. Δηλαδή, μια χώρα, εάν έχει δυσκολίε, θα πρέπει να ε, εξετάζεται κατά πόσο σεβάστηκε τους κανόνες, όχι αν κάποιον έχει παραβιάσει. Επίσης, ο κώδικας των κανόνων θα πρέπει να βασίζεται σε κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Κριτήρια τα οποία γράφεται να υπάρχουν σε αυτόν τον κώδικα της ε, σύγκλησης και να είναι ξεκάθαρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει τη λογική ότι οι πληρωμές και οι επιδοτήσεις για τις υποδομές θα πρέπει να υπόκεινται στο κατά πόσο είναι διαθέσιμα τα κονδύλια. Αυτή η προϋπόθεση της διαθεσιμότητας των κονδυλίων έχει διαγραφεί από τους συνεισηγητές. Πώς θα ξεκινούν ε, οι πληρωμές όμως αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, αν δεν είναι διαθέσιμες. Εγώ καλωσορίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι ε, προφανώς για να γίνουν πληρωμές πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο χρήμα. Ε, επίσης υπάρχει και η ιδέα του μηχανισμού ασφάλισης. Αυτό ήταν κάτι το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο όταν συζητήσαμε για την έκθεση αυτή και δεν υπήρξε καμία πλειοψηφία. Η συμμόρφωση υπάρχει. Το βλέπετε. Δεν είναι κάτι που λείπει. Λοιπόν, Μπέρντ, διόρθωσαν οι δύο συνάδελφοι. Κύριε Μπέγκε, πραγματικά σας εκτιμώ προσωπικά, αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει πουθενά η υπογραφή του ΕΛΚ. Αναγνωρίζω όμως ε, την υπογραφή των ε, σοσιαλδημοκρατών. Να σας πω γιατί είπα ότι είναι μια έκθεση ψευδής. Μας λέει ότι έχουμε ένα μηχανισμό επενδύσεων για μεγάλους ασύμετρους κρατασμούς, Αλλά η αιτιολόγηση είναι η οικονομική κρίση, η οποία ήταν ξεκαθαρά συμμετρικός κρατασμός. Επηρέασε αρνητικά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπήρξε κάποια ασύμμετρία. Το ότι εδώ πέρα μιλάμε για ασύμετρο σοκ και στα εκτιμώντας μάλιστα αναφέρεται ρητός η οικονομική κρίση, είναι ψευδές γιατί ε, ακριβώς έχουμε την πολιτική συνοχής ε, και εκεί έχουμε χρησιμοποιήσει αυτήν την αιτιολόγηση. Αλλά η οικονομική κρίση δεν ήταν κάτι τέτοιο, δεν ήταν ασύμετρος κραδασμός. Καλό είναι λοιπόν να ορίσουμε κάπου και να, να δούμε τον ορισμό του ασύμετρου σοκ. Επίσης, είναι κατά της οικονομίας της αγοράς γιατί δεν θα υπάρχει ένας μηχανισμός των επιτοκίων, αντιθέτως θα υπάρχει επιδότηση των επιτοκίων. Μιλάμε για κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία γιατί μιλάμε για αυτοματισμό και δεν υπάρχει καν η πρόθεση να μιλήσουμε για την αποδοτικότητα των επενδύσεων. Αρκεί μόνο να δώσουμε λεφτά χωρίς να δούμε εάν θα είναι κερδοφόρες αυτές οι επενδύσεις. Αυτό δεν έχει ούτε σχέση με η οικονομία της αγοράς. Επίσης δεν συμφωνώ με τον κύριο Μπέγκε όταν είπε και, είπε και η κυρία Μπερές κάτι ανάλογο ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας μηχανισμός ενεργοποίησης τον οποίο έχουμε σκεφτεί προσεκτικά. Αντιθέτως, αν δούμε την ε, ανεργία τότε το θέμα μας δεν είναι αντίδραση στο σοκ, αλλά η δυνατότητα αντίδρασης μιας οικονομίας. Και αν είναι ευέλικτη περισσότερο ή λιγότερο, σημαίνει ότι μια αγορά, μια ε, χώρα, μια οικονομία με πιο ευέλικτη αγορά εργασίας θα αντιμετωπίσει καλύτερα την κρίση σε σχέση με μια χώρα η οποία είναι πιο ε, άκαμπτη σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, ο μηχανισμό αυτό θα απευθύνεται σε αυτέ τι χώρε οι οποίε δεν έχουν κάνει τι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει που θα έπρεπε. Δηλαδή, εδώ πέρα δημιουργούμε λάθο κίνητρα. Και τελευταία παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, προφανώ δεν έχουμε σκεφτεί ποια είναι η σχέση μεταξύ τη προώθηση δημοσίων επενδύσεων που υποτίθεται επίση θα έπρεπε να έχουν μια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία που επίση δεν έχει καθοριστεί και των ε, επενδύσεων των ιδιωτικών που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και εδώ πέρα θα δημιουργήσουμε ένα φαινόμενο crowding out, θα διώξουμε δηλαδή ε, επενδύσεις. Έχουμε λοιπόν ένα μέσο που είναι κατά της ε, ελεύθερης αγοράς και είναι ψευδές. Γι' αυτό τα είπα αυτά. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να είναι σοσιαλιστικό, γιατί ε, με τη λογική σας το Δέλτα Νιτάφ είναι σοσιαλιστικό, η ΕΠΑ είναι σοσιαλιστική χώρα και όλες οι χώρες που έχουν αυτόματο σταθεροποιηθεί είναι σοσιαλιστικές. Ζούμε σε κόσμο σοσιαλιστικό λοιπόν, χωρίς να το ξέρουμε. Μα, μα κάτι μάθαμε και σήμερα. Λοιπόν, Ούρμα Σπάιτ από την Άλντε, απουσιάζει ο Ραμόν Τρεμόσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς. Και σε σχέση με αυτά που είπα προηγουμένως στην προηγούμενη συζήτηση, εμείς κάνουμε μια συζήτηση λογική ε, στους φιλελευθέρους. Όπως ξέρετε έχουμε διάφορες τάσεις ε, από διάφορες χώρες προερχόμενοι και διαφορετικούς πολιτισμούς. Έχουμε και διαφορετικές απόψεις για κάποια θέματα. Ε, ο συνάδελφος Μούρες, αν το είπε προηγουμένως, θα πρέπει να συζητήσουμε και τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Υπό ποια ανένεια. Η έκθεση αυτή ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και κάποιο καταμερισμό κινδύνου και περιορισμό κινδύνου, μείωση. Αυτό είναι το πλαίσιο το γενικότερο. Πολλά μέλη της ομάδας μου καταλαβαίνουν ότι πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στις διαφορετικές μεταφορ... μεταρρυθμίσεις συγγνώμη, και τη συμμόρφωση στο σύμφωνο σταθερότητα. σταθερότητας. Να σας εξηγήσω κάτι. Μπορεί να θυμάστε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από λίγα χρόνια ο πρόεδρος ομάδα, δι, ε, Ομπάμα διέσωσε τη General Motors που είναι αυτοκινητοβιομηχανία. City of Detroit. Αλλά δεν διέσωσε ο πρόεδρος Ομπάμα την πόλη του Detroit. Γιατί στο τέλος του 19 στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ε, σφυριλατούσαν την ένωση τους ε, έλεγαν θα έχουμε ένα μοσπονδιακό χρέος. Ε, συμφώνησαν λοιπόν όταν στείναν αυτό το σύστημα ότι δεν πρόκειται να ε, σώνουν με δημόσια χρήματα ε, πόλεις και πολιτείες. Άρα όταν υπάρχει αυτό το θέμα της αιρεσιμότητας, υπάρχει αυτό το στοιχείο. Δύο λεπτά και δεν τα ξεπερνάω, όπως και την περασμένη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, for the Greens, Ο Γιώργη Σολέ από τους Πρεσίνους, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την αδειά σα ε, θα πάρω και τα δύο λεπτά του συναδέλφου του κυρίου Λαμπέρτ. Είναι επιχορήγηση, δάνειο, τι είναι. Επιδότηση. Ε, είναι μια χάρη, χάρη από τον συνάδελφο. Ε, στην υπηρεσία του λαού. Mm. Ήδη 20 δευτερόλεπτα πέρασαν όμως. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε πέντε σημεία το πρώτο φορά το μέγεθο και εμεί θεωρούμε ότι 30 δισεκατομμύρια για την περίοδο 21-27 είναι λίγα και δεν επαρκούν. Εάν ο στόχος είναι να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μέσο να αντιμετωπίσει τους ασύμετρου κραδασμού. άρα προτείνουμε το επίπεδο να είναι τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ τη Ευρωζώνης. 120 δισεκατομμύρια δηλαδή. Που σημαίνει ε, πάλι το διπλάσιο από αυτό που προτείνουν οι συνεισήγητες στην τροπολογία 19. Επιπλέον, είμαστε υπέρ ε, του να προσθεθούν ε, ή να δοθούν επιχορηγήσεις αντί για δάνεια, καθώς θα έχουν περισσότερο σταθεροποιητικό χαρακτήρα. Δεύτερον, για την αιρεσιμότητα, πέρα από τη συμμόρφωση με του ουσιονομικούς κανόνες, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να μπουν κάποιοι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί όροι για την επιλεξιμότητα, παραδείγματο χάρη η επίτευξη των στόχων του 2020. Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου. Τρίτον, για τους δείκτες θεωρούμε ότι οι δείκτες ε, που θα χρησιμοποιηθούν ως ε, κριτήριο θα πρέπει ακριβώς να τους επεξεργαστούμε. Το να έχουμε δύο σωρευτικές ε, συνθήκες είναι πολύ περιοριστικές, ειδικά για τις χώρες που είχαν τα τελευταία 16 τρίμηνα τεράστια ανεργία. Για μας ένας όρος αρκεί για να υπάρχει πρόσβαση στο μέσο. Ε, θα πρέπει να αποκλείσουμε αλλιώς ε, κράτη-μέλη ε, τα κράτη-μέλη με ανεργία πάνω από το όρο της Ένωσης δεν θα πρέπει να πληρούν τους δύο όρους. Κατόπιν, για την φύση των επενδύσεων, βεβαίως η ομάδα μας θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρασίνισμα και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να μπουν και κάποια κριτήρια κοινωνικά και απασχόλησης. Και τέλος, για το δημόσιο χρέος θεωρούμε ότι τα ποσά που παρέχει το μέσο αυτό στα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξαιρούνται από τους υπολογισμούς δημοσίου χρέους. με το σκεπτικό ότι θα πάνε σε επενδύσεις για δημοσίες υποδομές ε, και αποτελούν ε, πρωτογενή σχηματισμό κεφαλαίου. Σας ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ υπάρχουν ομιλητές. Ε? Όχι. Η FDD δεν βλέπω. Η ΕΝΕΦ. Ο κ. Τζάνι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ συνοπτικά. θα Πρέπει να δούμε τα σημεία της πρότασης αυτής, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι πρόταση που θα λύσει προβλήματα στην Ευρωζώνη. Μου φαίνεται ότι είναι μια από τις πολλωστές, πολλαπλές απόπειρες που έχουν γίνει στο παρελθόν να λύσουμε ένα πρόβλημα διαρθρωτικό. Να αντιμετωπίσουμε με μια σπιρίνη όγκο, ε, καρκίνο. Τρία στοιχεία σημαντικά. Αυτό που είπε και ο συνάδελφος Λούκε, ότι ένα εργαλείο αυτής, αυτού, αυτής της φύσης δεν μπορεί να απορροφήσει τα συμμετρικά σοκ. Όμως δεν μπορεί να απορροφήσει και δεν μπόρεσαν και τα ανάλογα να απορροφήσουν ε, το σοκ της μεγάλης κρίσης, που δεν ήταν ε, συμμετρικό. Ήταν κάτι που έπληξε ολόκληρη την Ήπειρο. Και έπειτα, για άλλη μια φορά, με ένα εργαλείο ε, χρηματοδοτικού χαρακτήρα προσπαθούμε να λύσουμε μέρος του προβλήματος πρόβλημα που σε μια χώρα κανονικών συνθήκων έπρεπε να επιλύεται με νοσματικές πολιτικές. Οι κεντρικές τράπεζες ε, στην εντολή τους ε, έχουν το καθήκον να παρακολουθούν το επίπεδο της απασχόλησης και να αντιδρούν όταν αυτό δεν είναι στο ύψος των προσδοκιών. Εμείς εδώ προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα με ένα ακόμα εργαλείο που είναι αναποτελεσματικό Επίσης, η αιρεσιμότητα. Το να συνδυάσουμε, να προβλέψουμε τέτοια αιρεσιμότητα για αυτό το εργαλείο θα το κάνει αναποτελεσματικό για άλλη μια φορά. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη θα διστάσουν, θα επιφυλαχθούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό. Ε, και επίσης προσπαθούμε να αυξήσουμε τις συνεισφορές των κατομελών, ιδίω αυτών που τα τελευταία χρόνια ε, προσπάθησαν να στηρίξουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους ζητάμε περισσότερο χρήμα για ένα εργαλείο που ε, αντικειμενικά δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα διαρθωτικά, τα δομικά προβλήματα της Ευρωζώνης σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε στο Catch Ο κύριος Καλουέ Σαμπών και ο κύριος Χιον Χώνας Ποιος άλλος? Καλβέσσεμπον. Με ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις ιδέες θέλω να αναφέρω για να μην καταχραστώ του χρόνου σας. Το πρώτο που με ενέπνευσε ε, η τοποθέτηση του, του κυρίου Λούκε για την Ευρώπη ολόκληρη και την Ευρωζώνη ήταν συμμετρικός κραδασμός η κρίση, αλλά εντός της Ευρωζώνης ήταν ασύμετρες οι συνέπειες και εκεί θα πρέπει εμείς να παρέμβουμε. Έλεγε ο συμπατριώτης μου, ο Ισπανός από την Άλντε, ε, ε, μίλησε για το Τιτρόιτ, αλλά ε, και η Καλιφόρνια όταν είχε καταχρεοκοπήσει ε, δέχτηκε βοήθεια. Ήρθε ένας ομοσπονδιακός ε, ελεγκτής και έγινε παρέμβαση μέχρι και για να αγοράζει μολύβια ο κυβερνήτης στην Καλιφόρνια. Και τελειώνω. Υπάρχει και η, ε, άποψη της απασχόλησης. Ακόμα και για δεοντολογικούς λόγους πρέπει να καταγγείλουμε το γελίο ποσό. Ξέρω ότι είναι γελίος ο προπολογισμό για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό έχουμε και γελίους προϋπολογισμούς επιμέρους. Αλλά να θεωρήσουμε ότι τα μισά όσα δόθηκαν στην Ιρλανδία στην τελευταία κρίση θα αποτελέσουν αυτόματο σταθεροποιητή για την επόμενη, ε, είναι γελίο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να το καταγγέλουμε μπορούμε. Ξέρω ότι έχετε ζητήσει να είναι αυτόματη η ενεργοποίηση. Εμένα με ανησυχούν και οι ε, κοινωνικές συνέπειες ε, στην ε, ζήτηση μπορούμε να παρεμβούμε ως εξής, να βελτιώσουμε ή να διευρύνουμε τους κοινωνικούς παράγοντες, δείκτες. Ας πούμε, όταν επιδεινώνεται συνεχώς η φτώχεια. Ευχαριστώ και συγχαίρω τους συζητητές. δικτες ας πάρα πολλά από τη δουλειά τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χώνας, σε ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι το σημαντικότερο στην πρόταση αυτή είναι ότι ο σταθεροποιητής θα πρέπει να είναι πραγματικά αυτόματο, όπω είπε και η Περβάν Το πρόβλημα όμω ποιο είναι, όταν το βάζει σε σύστημα ε, εγγύηση ε, των επενδύσεων, οι επενδύσει τους ε, από τη φύση τους έχουν περίοδο ρήμανσης πολύ μακρύτερο. Ετοιμάζεται ένα σχέδιο, μελετάτε, υλοποιείτε και τελικά έρχεται η επένδυση χαιρετίσματα ε, για τον αυτόματο χαρακτήρα αν το προσανατολίσουμε στις επενδύσεις. Διότι προφανώς οποιαδήποτε σύστημα εγγύησης επενδύσεων θα έχει μια χρόνο καθυστέρηση από τη στιγμή που ενεργοποιείται μέχρι τη στιγμή που επενδύεται ε, το χρήμα αυτό. Το είπαν και οι συνάδελφοι προηγουμένω, οι Σοσιαλιστέ και οι δημοκράτες ότι για να εγγυηθούμε αυτό τον αυτόματο χαρακτήρα καλό θα ήταν να μην χρηματοδοτούμε τις επενδύσεις αλλά την κατανάλωση που αυτό κάνει αυτόματο το σύστημα. Και αυτό θέλουμε εμείς να μεταρρυθμίσουμε ε, το σύστημα σε ένα σύστημα προστασίας της ανεργίας εξού και η αυτοματοποίηση του συστηματο. Αν από την άλλη θέλουμε να εξακολουθήσουμε να έχουμε ένα σύστημα που θα σταθεροποιεί βάσει των επενδύσεων, ε, τότε θα έπρεπε να διατηρήσουμε στο πρόγραμμα EU Invest ή e Invest EU κάποια αντικυκλικά προφίλ χρησιμοποιώντας την εγγύηση ε, τους πολλαπλασιαστές έτσι ώστε το EU Invest να ασχολείται με τις επενδύσεις που κατά τα άλλα είναι ιδιωτικές επενδύσεις για να κινητοποιούνται πιο γρήγορα και από την άλλη αυτόματο σταθεροποιητής να προορίζεται στην κατανάλωση και μόνο για να έχουμε αυτή την αντικυκλική ε, συνέπεια και λειτουργία που φιλοδοξούμε. Ευχαριστώ, Jean Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους δύο συνεισηγητές μας που εδώ και τρία χρόνια με ιδιαίτερη ε, αποφασιστικότητα επιδιώκουν να ετοιμάσουν μια τέτοια, αυτή την πρόταση. Είναι άοκνες προσπάθειές τους και η επιμονή τους με εκπλήσει, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της δεν μας ε, ικανοποίησε πλήρω. Για άλλη μια φορά ε, προτείνεται ένα εργαλείο που δεν είναι στο ύψος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, το κοινό νόμισμα, η κοινή νομισματική πολιτική δεν συνδυάζεται με τις πολλαπλές εθνικές πολιτικές. Αυτό που εδώ συζητούμε είναι η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης η οποία παραμένει πολύ εύθραυστη με σοβαρούς κινδύνους και τα 30 δις δεν είναι στο ύψος των ε, κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσουμε αύριο. 30 δις είναι πίνατς, είναι σαχλαμάρες, τίποτα. Ε, πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι με τις πολιτικές μας για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Συγχαίρω λοιπόν τους δύο συνεισηγητές, έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά εδώ απευθύνουμε έκκληση στους αρχηγούς ε, κρατών και κυβερνήσεων για να αλλάξουν λίγο το software που χρησιμοποιούν. Ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι ότι μας έχουν μείνει μόλις πέντε λεπτά, οπότε δεν θα μιλήσω γιατί με κάλυψε ο συνάδελφος. Όσον αφορά λοιπόν την αποτελεσματικότητα, την τεχνική πτυχή της δυνατότητας να απορροφηθούν ασύμμετροι κραδασμοί, νομίζω ότι έχετε δίκιο. Ε, το επίδομα ανεργίας ε, είναι ο πραγματικός αυτόματος ε, σταθεροποιητής. Και μετά μπορούμε βεβαίως να μιλήσουμε για σήμανση κτλ. Αλλά δεν είναι καθόλου ασύμβατο αυτό αλλά θα ήθελα οι συνεισηγητές να σκεφτούν ε, ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για να δούμε τον στόχο που φαίνεται να έχουμε κοινό. Κομισιόν, σύντομα όμως, γιατί μετά θα πρέπει να δώσουμε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους δύο συνεισηγητές για την διαφωτισμένη τους ε, προσέγγιση προς την πρωτοβουλία αυτή της Κομισιόν έχουν αντιληφθεί το τι διακυβεύεται. Αυτό είναι το πρώτο συγκεκριμένο βήμα των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων για έναν μηχανισμό συλλογική αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν ασύμετρους κραδασμούς καθώς έχουν, ε, δεν έχουν πλέον την δυνατότητα που τους παρήχε η συναλλαγματική ισοτιμία. Πρόκειται δηλαδή για κάτι το θα βοηθήσει χώρε οι οποίε έχουν χρηστή διαχείριση όταν αντιμετωπίζουν κάτι εκτό του ελέγχου του πριν βρεθούν σε ανάγκη να χρειαστούν ένα δομημένο πρόγραμμα βοήθεια. Αυτό είναι ο στόχο. Θα συμβούν αυτοί οι κρατασμοί, έχουν ξανασυμβεί, καταραίουν ε, συχνά και οι τιμέ των ακινήτων. Ε, έχουμε ε, άλλε χώρε στην Ανατολική Ευρώπη που βρίσκονται σε μια δύσκολη γειτονιά Πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε και το σχέδιο έκθεσης ορίζει, θα λέγαμε, το πλαίσιο και για αυτό το οποίο είπατε για το επίδομα της ανεργίας νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πλέον ε, διαδίδεται στις πρωτεύουσες ε, και υπάρχουν κάποιες πρώτες ε, κρούσεις στο Συμβουλίο Κομισιόν. Οπωσδήποτε θα το δει το θέμα επικοδομητικά. Θα προσπαθήσουμε να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση Πρέπει να συμβαστούμε τη νομική βάση, να αποφύγουμε το να εστιάσει το θέμα στα επιδόματα ανεργίας ε, και να μην επηρεάσει έτσι τον αυτοματισμό και την γρήγορη χρήση και να μην μπουν όροι ε, στα εθνικά συστήματα επιδόματος ανεργίας. Αλλά υπ' αυτούς τους όρους θα ακολουθήσουμε το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη στην κατεύθυνση που αυτά θέλουν. Ε, σύντομα για το μέγεθος του προϋπολογισμού. Δεν είναι αυτό το μόνο μέσο που έχουμε για την αντιμετώπιση της κρίσης αφορά τη σταθεροποίηση των δημοσίων επενδύσεων πριν ε, πληγεί μια χώρα από την κρίση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στο ΠΔΠ αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούσε να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο στην σταθεροποίηση μέχρι και ενός 10% των δημοσίων επενδύσεων. Είναι μέρος της λύσης και είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση που πρέπει να πάμε. Και τέλος, Καλωσορίζουμε τις ε, δηλώσεις ε, της κυρίας Μπερές για τους όρους ενεργοποίησης, ε, για τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Πρέπει ο μηχανισμός αυτός να είναι στόχευμένος σε αυτούς οι οποίοι το αξίζουν στις χώρες με την καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση, οπότε θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προσπάθειες του να προωθήσει αυτήν την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Ποιο θέλει να ξεκινήσει, ο κύριο Μπέγκε. Ναι, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος ε, Λούκε έχει ε, δίκιο, δεν ήταν ενωμένη ομάδα του ΕΛΚ, αλλά κατά πλειοψηφία ήταν ε, στο πλευρό μου και χάρηκα γιατί αυτό ήταν το σωστό. Κοιτάξτε, όταν μιλάτε για ψεύδι, εγώ ευθυγραμμίζομαι με το ΔΕΛΤΑ με τον Κλάους Ρέγκλινγκ που είναι αναμφισβήτητα ειδικό και με τον καθηγητή Φιούστ του Ινστιτούτου του Μονάχου, με τον κύριο Ντιμάουρο, δηλαδή με ε, ειδικού εγνωσμένου ε, κύρους. Δεν είμαι τόσο ειδικό στα οικονομικά, αλλά θυμάμαι ότι τα οικονομικά δεν είναι θετική επιστήμη, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής. Ζίγκριτ Μορεσάν, δείτε τους ορισμού. Λέει ότι υιοθετείται με βάση την τακτική νομοθετική διαδικασία. Πρέπει να μπει, ναι, το διατυπώσαμε έτσι, υπάρχει μια σχέση και νομίζω ευχαρίστω να το ξεκαθαρίσουμε. Ακριβώς ε, ορίσαμε ως ενεργοποιητή το επίπεδο της ανεργίας, ε, το, γιατί το Συμβούλιο είπε ότι εάν θέλουμε να έχουμε έναν αυτόματο ενεργοποιητή, αυτός είναι ο καλύτερος και ο σαφέστερος. Αλλιώς μπορούμε να διατυπώσουμε ε, δέκα πτυχές ε, και δεν θα λειτουργεί τίποτα. Δεύτερον, να ξεκαθαρίσω και πάλι, αυτό το οποίο κάνουμε εμείς ε, εδώ πέρα, με τις τροπολογίες, δεν είναι, δεν σημαίνει ότι δίνουμε εξοδότηση λευκό για μια ασφάλιση ανεργίας. Διακόπτεται η διερμηνία, ρωτάει ο κύριος Ε, πρέπει να σταματήσει η διερμηνία εδώ, τελειώνει η διερμηνία με βάση το πρόγραμμα. Οι διερμηνείς έχουν και άλλη συνεδρία στη συνέχεια. Which was presented also from Minister Scholz. Um, yes, you may discuss it, but it was something we at this point didn't want to have as amendments to go in what direction because there we have different differences